Bene, cominciamo i nostri lavori del pomeriggio. Συνεχίζουμε λοιπόν τις εργασίες μας. Ξεκινάμε με το επόμενο σημείο της διατάξεως, συμπληρωματικό πρόγραμμα έρευνας για το έργο ΙΤΕΡ, με το λόγο έχει ο συνάδελφος ΡΕΜΕΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα φροντίσω να είμαι σύντομος ε, και σαφής. Νομίζω ότι το πρόγραμμα ITER έχει ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία, διότι η σχάση έχει, η σύνδεξη έχει μεγάλη σημασία στον τομέα της ε, ηλεκτρικής ενέργειας και την σχετική παραγωγή και είναι ε, μια διαδικασία ε, θετική για το περιβάλλον, φιλική προς το περιβάλλον. Το πρόγραμμα το οποίο όμως προτείνει η Κομισιόν δεν είναι κατάλληλο για την ε, εφαρμογή του. Νομίζω ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μια διαφορετική χρηματοδότηση δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι και χώρα υποδοχής θα πρέπει να αποστείλει ε, ένα σαφές μήνυμα ότι θα συνεχίσει να στηρίζει το έργο ITER και το Κοινοβούλιο θα μπορεί να έχει με αυτόν τον τρόπο έναν καλύτερο έλεγχο στις, στον χρηματοδότηση αλλά και στον προπολογισμό του ΙΤΕΡ. Γι' αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί στο πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχουν λεπτομέρειες που θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τους κοιόδης ηγητές. Έχω ε, συνεργαστεί με πολλούς εξ αυτών στο παρελθόν και σας ευχαριστώ εκ των προτείνων και προσβλέπω στις γνώμες σας και στα σχόλιά σας. Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Βινταλ Κουάντρες έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ με τη θέση του κυρίου Ρέμεκ. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Τι θέλουμε να κάνουμε. Να εγγυηθούμε τη χρηματοδότηση του ΙΤΕΡ. Και γι' αυτό λέγουν ορισμένοι. Καλύτερα να το κάνουμε αυτό στα πλαίσια του πολιετούς. Άλλοι λέγουν, όπως η Επιτροπή Φερρυπίν, καλύτερα να εγγυηθούμε τη χρηματοδότηση εκτός του πολιετούς χρηματοδοτικού πλαισίου. Και περιμένουμε από βάση του Συμβουλίου. Εάν όμως χρειαστεί να αυξηθούν τα κονδύλια που δίδονται στο ΙΤΕΡ, πράγμα το οποίο γίνεται γιατί πάντα υπερβαίνουμε τα ποσά τα οποία δίδονται. Εάν το έχουμε μέσα στο πλαίσιο, θα πρέπει να γίνεται ανακατανομή των κονδυλίων εντός του πλαισίου με όλα τα συναφή πολιτικά προβλήματα. Εάν είμαστε εκτός πλαισίου, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δώσουν απευθεία συμπληρωματικά κονδύλια. Και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα κράτη-μέλη θα το κάνουν αυτό χωρίς περαιτέρω δυσκολίες και συζητήσεις. Και οι δύο εναλλακτικέ λύσεις λοιπόν είναι, εναλλακ... είναι προβληματικές αν χρειαστούν συμπληρωματικά χρήματα. Εμείς ως Κοινοβούλιο τι έχουμε να πούμε. Αν βρίσκεται το ίτερ εντός του πλαισίου θα είμαστε από αυτούς θα λάβουν την απόφαση. Εάν βγει, απλώς θα ζητηθεί η άποψή μας και τίποτα περισσότερο. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε και ο κύριος Ρέμεκ. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε να παραμείνει το ίτερ εντός του πολιετούς χρηματοδοτικού πλαισίου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκλάντε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κάτι που πρέπει να τονίζετε διαρκώς είναι ότι αυτό το ITER είναι τεχνολογία απολύτως διαφορετική από αυτή της χάσης που χρησιμοποιείται τώρα για την παραγωγή ενέργειας. Σημαντικό διότι η σύνδεξη δεν έχει φτάσει ακόμα και πόρο απέχει από το σημείο να είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμη στην Ευρώπη. Ωστόσο να μην χάσουμε την ενδεχόμενη ευκαιρία στο μέλλον, γιατί αυτή θα μπορεί στατεύσει και το κλίμα. Στην τεχνολογία αυτή, εάν κάποτε εφαρμοστεί, το ενδιαφέρον είναι ότι είναι πολύ περιορισμένα τα, κατάλοιπα, τα ραδιενεργά κατάλοιπα τους, αλλά και στην ημιζωή τους, δηλαδή είναι της τάξης των 100 ετών. Κοστίζει πολύ ή λίγο θα μας κοστίσει πολύ εάν βγούμε από το πρόγραμμα αυτό. Υπάρχουν υποπροϊόντα αυτής της έρευνας που είναι χρήσιμα για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Εάν εξετάσουμε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τι τεχνογνωσία αποκτούν με τεχνικές συγκολήσεων κλπ. παράγοντας προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην έρευνα αυτή, θα δούμε ότι το όφελος είναι πολύ μεγάλο. Τα χρήματα βέβαια είναι το κέριο σημείο, τα κονδύλια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ενταχθεί ξανά στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ωστόσο να αποφύγουμε ένα πράγμα. Να βρεθούμε ξανά στο δίλημα να χρειαστεί να περικόψουμε σημαντικά τα κονδύλια του Twitter εποφελία άλλων προγραμμάτων. Ούτε θα είναι βέβαια εύκολο εάν εκτοξευθούν ε, οι δαπάνες για το θέμα αυτό, να φέρουμε αντιρρήσει σε κάτι τέτοιο. Ε, κατά τα λοιπά συμφωνώ με την προσέγγιση του κύριου Ρέμεκ. Ο κύριος Ρούμπικ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το πρόβλημα έχει πολλές πτυχές. Θα το βάλουμε στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, δηλαδή στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και κατά πόσο θίγεται τότε ο ορίζον 2020. Εάν το αφήσουμε απέξω το ΙΤΕΡ από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και αναμένουμε συμφωνία στο επίπεδο των Υπουργών, τότε θα είναι επιπρόσθετο πακέτο για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ή θα είναι καθαρά διακυβερνητική συμφωνία. Και τι θα γίνει τότε με την αδυναμία καταγγελίας της σύμβασης την οποία ήδη έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ θεώρησα πάντοτε ότι πρέπει να πούμε ναι, έχει καλώ. Πάκτα sunt σερβάντα. δηλαδή τα συμφωνηθέντα, οι συμβάσει πρέπει να τηρούνται. Αυτό είναι άλλωστε και η ευνοϊκότερη παραλλαγή. Δηλαδή πρέπει να παραμείνουν τα κονδύλια αυτά, τα συμφωνηθέντα κονδύλια στο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Και αν δεν συμβεί αυτό, πρέπει να υποβάλει η Κομισιόν πρόταση για το πώ, ποια μορφή μπορεί να λάβει μια ενδεχόμενη διακυβερνητική συμφωνία, έτσι ώστε να ε, σέβεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υποχρεώσεις που είχε ήδη αναλάβει. Ο κύριος Ρόιλ. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Ρέμεκ και τον υποστηρίζω και στους στόχους που προτείνει. Έχουμε κατά, κατ' επανάληψη συζητήσει περί της σκοπιμότητας των κοντιλίων αυτών, του μεγέθους των κτλ ως Κοινοβούλιο έχουμε πει ότι αποδίδουμε μεγάλη αξία στην ορθή οργάνωση και στη σωστή χρηματοδοτική υποστήριξη. Από την άλλη όμως, και επίσης σωστά το έχουμε τονίσει, πρόκειται για ένα έργο το οποίο έχει τεράστιες επιπτώσεις στην ενέργεια, στην οικονομία, στην έρευνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί και με πολλούς άλλους σημαντικούς παίκτες στον κόσμο Εάν θέλει να συνεχίσει να παίζει πρωτοπόρο ρόλο ε, στην προσπάθεια αυτή, πρέπει ε, να επιμείνει, πρέπει να αντέξει το ρόλο αυτό. Βρίσκω ότι είναι ύψη τη σημασίας η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έργο. Σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, συμφωνώ με τους άλλους συναδέλφους και δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτε. Εν τέλει, συνοψίζω λέγοντας ότι θα υποστηρίξω ευχαριστώ τον κύριο Ρέμεκ. Το λόγο έχει Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλό από μεσήμερο. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ ενώπιό σα, γιατί είναι η πρώτη φορά που σας ομιλώ ως ε, Γενικός διευθυντή, στην ε, Αρμόδια Διεύθυνση και έρευνας. Το ITER είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά την συνεργασία με 7 εταίρους και φέρει τον τίτλο «Ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης» και έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα της βιομηχανίας η Κομισιόν έχει προτείνει ένα συμπληρωματικό ερευνητικό πρόγραμμα εκτός του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου όπου θεωρείται ότι είναι και το αποτελεσματικότερο μέσο για τη χρηματοδότηση ενός παρόμοιου προγράμματος όπως το ITER. Γιατί, διότι θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε μια δέσμευση των κρατών μελών απέναντι στο πρόγραμμα αποφεύγοντας ε, ε, την μεταφορά σε άλλες γραμμές του προπολογισμού το πρόγραμμα και δεν θέλω να μακρηγορήσω αλλά η πρόοδος ε, είναι καλή και Η κατασκευή των κτηρίων προχωράει. Και όλα τα σχετικά προοδεύουν ικανοποιητικά. Έχει συσταθεί μια ομάδα, ήτερ. αλλά και κάποιες οργανώσεις ε, που ασχολούνται με το θέμα της ε, σύνδεξης. Ε, σημειώθηκαν ε, τα σχόλιά σας και αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν για το κατά πόσο το προβλήμα του ΙΤΕΡ θα βρίσκεται εντός ή εκτός του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. και όπως είπαν πολλά μέλη δεν ε, ε, θα χρησιμοποιούν για άλλους λόγους ε, τα κονδύλια του Twitter. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα, πάντως αν θέλετε μπορώ να απαντήσω σε ανεχόμενες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε την Κομισιόν. Προτού να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Ρέμι, να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο Έλερ, που είχε κάποιες δυσκολίες να φτάσει στη συνεδρίασή μας καιρός. Παρακαλώ. Um, <clears throat> zum, um... Για το θέμα Ίτερ, πριν από τα Χριστούγεννα, καταλήξαμε σε ένα συμβιβασμό και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν εξήγησε ότι δεν αφορά αυτό τον ορίζοντα 2020. Για τον πυλώνα 1α και τον ορίζοντα 2020, ωστόσο, η διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο είναι, δείχνει μια διαφορετική εικόνα. Για το Συμβούλιο βρίσκω ότι είναι αυτονόητο ότι θα χρηματοδοτήσει το ίτερ. Στον πυλώνα 1α δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια για τη χρηματοδότησή του. Έτσι λοιπόν με εκπλήσει λίγο αυτή η αισιοδοξία που διαπιστώνω ότι δήθεν το πρόβλημα κοντεύει να επιληθεί, ενώ ο τριμερής διάλογος και οι σχετικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο δείχνουν κάτι άλλο. Αυτό που θέλω τώρα να επισημάνω είναι ότι το Κοινοβούλιο, ναι μεν υποστήριξε τον προπολογισμό για το 2013, άλλωστε εδώ και πολλά χρόνια το Κοινοβούλιο προσφέρει υποστήριξη στο έργο ΙΤΕΡ, αλλά ο τρόπος της διάθεσης των κονδυλίων καθώς και τα θέματα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα παραμένουν. Και μάλιστα η θέση αυτή υπήρξε διακομματική. Για να προωθήσουμε το έργο αυτό, παραγωνίσαμε κάπως τις επιφυλάξεις αυτές, τις βγάλαμε λίγο από την παρένθεση, αλλά δεν έχουν απαλληφθεί. Τώρα υπάρχει και ένα ερώτημα που μέχρι τώρα δεν έχει απαντηθεί ποτέ μέχρι τώρα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει δημοσιονομικά τι θα γίνει εάν δεν συνεχίσουμε το ε, πρόγραμμα ITER. Βλέπουμε κάθε φορά μονάχα τις ενδοευρωπαϊκές συμβάσεις. Όμως τι γίνεται, εάν διαβάσει κανείς προσεκτικά τις συμβάσεις, θα δει ότι στο διεθνές πλαίσιο δεν είμαστε σε θέση να αποχωρήσουμε γιατί θα αναγκαστούμε να πληρώσουμε τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια ευρώ στην περίπτωση αυτή. Αυτό το ερώτημα έχει μείνει πάντα ανοιχτό μέχρι τώρα. Εάν κάτι τέτοιο θα επιβαρύνει τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, τον πυλώνα 1α. Έτσι λοιπόν το ερώτημα αυτό εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτό. Πάνω από μια διετία θέτουμε την ερώτηση αυτή και θα θέλαμε να ακούσουμε από την Κομισιόν και τις αρμόδιες υπηρεσίες πώς έχει η απάντηση. Γιατί για λόγους σαφήνειας του προϋπολογισμού θα πρέπει αυτό το ερώτημα καταρχήν να απαντηθεί. Ωραία, εάν η Κομισιόν θέλει να προσθέσει κάτι και μετά δώσουμε το λόγο στον κύριο Ρέμεκα. Όπως είπε ο κύριος Έλλερ, αυτό είναι μέρος διεθνούς συμφωνίας και όπως ελέγχθηκε προηγουμένως, νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρώπη να τιμά τις διεθνείς της δεσμεύσεις. Δεν ξέρω, λοιπόν, τι θα μπορούσαμε να προβλέψουμε για να αποσυρθούμε. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Δεν, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση νομίζω. Απ' την άλλη, το προηγούμενο έτος έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες συγκράτησης και περιορισμού του κόστους. Και έχουν και φέτος προβλεφθεί συγκεκριμένα μέτρα για να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. So, just to translate that to, to the simple mind of, of a parliamentarian. Σέλερ, στο απλοϊκό ίσω μυαλό ενό Ευρωβουλευτού αυτό σημαίνει ότι ούτω ή άλλω θα κληθούμε να πληρώσουμε. Είτε δηλαδή συμμετέχουμε κατά το μέρο μα, δηλαδή υλοποιούμε αυτά που έχουμε αναλάβει, είτε καλούμαστε να πληρώσουμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Προσπαθώ να το μεταφράσω σε απλά λόγια, διότι είναι διεθνεί υποχρεώσει που έχουμε αναλάβει. Στην περίπτωση όπου δεν εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει, τότε καλούμε θα να πληρώσουμε, έτσι δεν είναι. Απάντηση της Κομισιόν. Με συγχωρείτε. Μια στιγμή λέει η, η πρόεδρος. Κύριε Γκλάντε εσείς. Εδώ θέλω κι εγώ να επιμείνω λίγο. Εγώ είχα εξηγήσει τότε στους συναδέλφους της ομάδας μου και τους το είχα καταστήσει ελκυστικό, είπα ότι αν δεν τηρήσουμε τις διεθνείς μας υποχρεώσεις θα πληρώσουμε 4,2 δισεκατομμύρια. Εάν δεν βγούμε τότε έχουμε περίπου 2 δισεκατομμύρια. Καλά λοιπόν εντάξει είπαν τότε αυτοί συν 2 δισεκατομμύρια αλλά τότε υποφελούμεθα από τα τεχνολογικά επιτεύγματα. Αν όμως έρθετε τώρα και μας ε, πείτε ότι όλα αυτά δεν έχουν απολύτως καμία αξία πληρώνουμε και τελείωσε. Ας ξεχάσουμε όλη την ιστορία αυτή περί δημοσιονομικών. Commissione, prego. Yes. Concerning the statement whether or not uh, Euratom, represented by the Commission, can withdraw the ITER. Μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι αν αποσυρθεί η Κομισιό δεν μπορεί να το κάνει μονομερός. Διότι υπάρχουν κυρώσεις κυρώσεις προς τους άλλους εταίρους. Εκτός από τις κυρώσεις την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Κατεκτήμηση το ποσό που αναφέρατε ε, είναι απλώς κατεκτήμηση. Δεν μπορούμε να το ε, επιβεβαιώσουμε, αλλά θα υποστούμε ποινικέ ρήτρε. Αλλά προ το παρόν τα ποσά δεν μπορούμε να τα επιβεβαιώσουμε. Ναι, για τα συμπεράσματα το λόγο ο εισηγητή. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χάρηκα πολύ που άκουσα τις απόψεις των συναδέλφων μου. Ιδιαίτερα διαφωτιστικές. Έχω και την γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, η οποία ανησυχεί ότι μεταφορά των χρηματοδοτήσεων σε άλλες γραμμές του προϋπολισμού μπορεί να μειώσει την ε, ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τεχνολογική καινοτομία και ανάπτυξη. Οι νέες τεχνολογίες συχνά βασίζονται σε μη αναμενόμενα αποτελέσματα της έρευνας. Χάρηκα πάντως που άκουσα τις ε, γνώμες σας, τις απόψεις σας. Δεν συμφωνούμε βέβαια πάντοτε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι στις επόμενες συναντήσεις μου με σκιώδεις συγητές και άλλα αρμόδια πρόσωπα θα καταλήξουμε σε αποδεκτούς συμβιβασμού, στοχεύοντας σε μια λύση που θα επιτρέψει την εφαρμογή του προγράμματος ITER. Ούτε τολμώ να διανοηθώ ότι μπορεί να εγκαταλείψουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Είναι. Υπενθυμίζω πως οι τροπολογίες ε, του προγράμματος ε, του και η εξέτασή του προβλέπεται για ε, τις 20 και 21 Φεβρουαρίου. Αυτή είναι η ημερομηνία για την εξέταση των τροπολογιών και την συζήτηση. Ε, προσπάθησα να μάθω αν μπορούν να φτάσουν νωρίτερα οι υπουργοί, αλλά δήλωσαν ότι δεν μπορούν να φτάσουν πριν από τις 17.00. Διακόπτουμε για 30 λεπτά τη συνεργασία μας. Παρακαλώ τους συναδέλφους να επιστρέψουν εγώ με τα χαράς να κάνω παρέα στους υπουργούς, αλλά ελπίζω να έχω και κάποιον συνάδελφο μαζί μου να υποδεχθούμε τους υπουργούς. Ευχαριστώ. Τα λέμε σε λίγο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τις εργασίες μας. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Αναφίβολα θα φτάσει και κάποιος ακόμα συνάδελφος. Περιμένουμε ακόμα μερικά λεπτά διότι έχουμε και κάποιους καθυστερημένους. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Ρίτσαρτ Μπράτον, Ιρλανδό Υπουργό, για θέματα εργασίας, επιχειρήσεων και καινοτομίας και τον κύριο Σον Σέρλοκ, που είναι υφυπουργό στο αυτό Υπουργείο και ασχολείται ιδιαίτερα με θέματα ενέργειας και καινοτομίας. Βρίσκονται εδώ εκπροσωπώντας την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που ανέλαβε κατά τη διάρκεια του Ιρλανδικού εξαμήνου. Σήμερα το πρωί είχαμε τον Υπουργό κύριο Πατ Ράμπιτ και σήμερα θα ολοκληρώσουμε την συνεδρία μας με την παρουσία του κύριου Ρίτσαρντ Μπράτον και του Σον Σέρλοκ, τους οποίους και ευχαριστούμε για την παρουσία τους. Θα του δώσουμε 30 λεπτά για την παρουσίαση. Θα δούμε πώς θα μοιράσουμε μεταξύ τους τον χρόνο και έπειτα θα ακολουθήσει συζήτηση με τους συναδέλφους και τα, ε, τα συμπεράσματα των κυρίων Υπουργών, τους οποίους ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά, που ήρθαν στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, Επιτροπής Ενέργειας, Βιομηχανίας και Έρευνας, μετά από την έναρξη των εργασιών το 2013. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μεγάλη τιμή και για μένα και το συνάδελφο Σεν Σέρλοξ. Είμαστε παρόντες, λάβουμε το λόγο στην Επιτροπή σας. Στη δεκαετία του 90 στην προηγούμενη μας Προεδρία δεν συμμετείχε στην διαδικασία συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σήμερα με ευχαρίστηση βλέπουμε πόσο έχουν αυξηθεί οι αρμοδιότητές σας και στα πλαίσια των ε, πρωτοβουλειών. Ο συνάδελφος ασχολείται με τα θέματα καινοτομία και έρευνα και εγώ με τα θέματα της ε, βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας. Προσπαθούμε τα θέματα που μας απασχολούν να τα χειριστούμε με, ο καθένας με τον τρόπο του ως Προεδρία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη και να μειώσουμε το άχθος για τις ε, ε, μικρομεσαίες επιτυχήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε τους ε, ιδρυτές δυνητικούς και τους παράγοντες των νέων επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουμε να τους δώσουμε τις καλύτερες δυνατές δυνατότητες που προσφέρουν για να δημιουργήσουν τις επιχειρήσεις τους. Χαιρετίζουμε την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σχέδιο δράσης επιχειρηματικότητα 2020 και υποστηρίζουμε τους στόχους της, κυρίως αυτούς που αφορούν την υποστήριξη και προώθηση των επιχειρηματιών και θα θέλαμε να επιστηρίξουμε περισσότερο την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη. Προβλέπουμε ε, επί αυτού του θέματος να συζητήσουμε στο άτυπο συμβούλιο επιχειρηματικότητας που θα γίνει το Μάιο και ελπίζουμε και εσείς θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε. Η ΜΜΕ όντως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ευρώπης και συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη της Ευρώπης. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε προτεραιότητα σε διάφορα μέτρα που θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση στις ε, δυνατότητες ε, για τις κρατικές προμήθειες και υποστήριξη της ε, συμφωνίας Κόσμε για την παροχή βοήθειας είναι κλειδί και θα το υποστηρίσουμε για τη διάρκεια της Προεδρία μας. Επίσης υποστηρίζουμε ε, τον ε, γενικό στόχο αυτού του προγράμματος και χαιρετίζουμε την διευκόλυνση ιδίων πόρων για τις ε, επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στη φάση της ανάπτυξης και την διευκόλυνση δανειοδότησης που θα δώσει, ε, που θα προσφέρει ρυθμίσεις ε, με τους ε, χρηματοπιστωτικούς μεσάζοντες για δάνεια για τις ΜΜΕ. Βεβαίως το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα αποτελέσει το πλαίσιο για το προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2014-2020 και τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για το πλαίσιο αυτό θα καθορίσουν τις προοπτικές που έχουμε για να προοδεύσουμε μεταξύ άλλων και στο πρόγραμμα COSME. Yeah. Όπως σας είπα, αυτό είναι μέρος του άτυπου Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας που θα λάβει η χώρα στο Δουβλίνο το Μάιο. Η εστίασή μας θα είναι στις ΜΜΕ ως φορέα ευρωπαϊκής ανάπτυξης και επιπροσθέτως η Επιτροπή θα συγκαλέσει και το φόρουμ χρηματοδότησης των ΜΜΕ στις 2 Μαΐου στο Δουβλίνο σε συνδυασμό με το δικό μας άτυπο συμβούλιο. Όπως ξέρετε θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η εποπτεία της αγοράς, πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση των ΜΜΕ στην χρηματοδότηση και σε αυτό το υψηλού επίπεδου φόρουμ θα συναντηθούν πρόεδροι, γενικοί γραμματείς ε, βιομηχανικών οργανώσεων, πιστοτικών ιδρυμάτων, τραπεζών, καθώς και ο Επίτροπος Ταγιάννη, ε, ευρωβουλευτές και εκπρόσωποι της Προεδρίας. Ο Επίτροπος θα μπορέσει να σας ενημερώσει εκ των υστέρων για τα συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξουμε. Όσον αφορά την βιομηχανία και τα θέματά τους. Όπως ξέρετε, η παγκοσμιοποίηση είναι μια μεγάλη πρόκληση για τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται διάφορες εταιρείες και γενικότερα οι βιομηχανίες. Η έκθεση του 2012 για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα τονίζει πόσο σημαντικές είναι ο ρόλος των παγκόσμιας αξίας ε, αλυσίδων για την βιομηχανία μας. Μία, και θα αναφέρω και θα τονίσω ιδιαίτερο την ε, σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια ενοποιημένη βιομηχανική πολιτική την εποχή της ε, παγκομισμιοποίησης. Υπάρχουν ε, νέες προοπτικές που, χρειάζεται, που απαιτούν να αλλάξουμε την προοπτική μας και να δημιουργήσουμε νέα δίκτυα και κόμβους για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις βιομηχανίες μας. Η δική μας Προεδρία θα συνεχίσει την ε, πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί σε θέματα μείωσης του βιομηχανικού κόστους από των ε, προγραμμάτων μείωσης του διοικητικού άχθους και θα προσπαθήσει να βοηθήσει όλες τις επιχειρήσεις. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν συμπεράσματα τα οποία θα καταλήξουμε μετά τον ε, ε, Συμβούλιο του Μαΐου και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας για να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτό το άχθος. Θα πρέπει να βρούμε νέους τρόπους για να μειώσουμε το διοικητικό αυτό των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να δούμε πού υπάρχουν προβλήματα και πώς μπορούμε να τα μειώσουμε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μία ευφυή νομοθεσία που θα μας βοηθήσει, κυρίως τις μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον που θα τους επιτρέψει να αναπτυχθούν και να ανθίσουν. Χαιρετίζουμε τις προτάσεις Επιτροπής σε σχέση με την πρωτοβουλία εξυγχρονισμού των κρατικών ενισχύσεων. Όπως ξέρουμε, οι στόχοι αυτής της διαδικασίας, κυρίω η ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνητη διαφάνεια προβλεψιμότητα και ορθολογισμό των διαδικασιών έχει ως στόχο να βελτιώσει τα πράγματα. Ε, αυτή η πρωτοβουλία εξυγχρονισμού των κρατικών ενισχύσεων έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Τη στιγμή κατά την οποία αντιμετωπίζουμε αυτή την οικονομική κρίση που θέλουμε να ξεπεράσουμε και θέλουμε να κάνουμε μια αγορά πιο δυνατή, πιο δυναμική και πιο ενοποιημένη. Θέλουμε στα ε, πλαίσια αυτών των πρωτοβουλειών να έχουμε ένα καθεστώς κρατικών ενισχύσεων πιο απλών, πιο σαφών και πιο ευέλικτων για να επωφεληθούν όλα τα κράτη-μέλη. Είμαι σίγουρος ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν τα κράτη-μέλη να έχουν πρόσβαση ακόμη και σε μικρότερες ενισχύσεις. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ενώ το καθεστώς αυτό είναι σημαντικό για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν για όλους ίσοι κανόνες πρόσβασης εντός της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει συγχρόνως η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι έτοιμη να ανταγωνιστεί με τρίτε χώρε για να κινητοποιήσει τι άμεσε ξένε επενδύσει τι οποίε χρειάζεται. Οι κρατικέ ενισχύσει επίση μπορεί να δοθούν από τρίτε χώρε σε επιχειρήσει και πιστεύουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συνεχίσει να το εξετάζει η Επιτροπή. Η Προεδρία μα θα προεδρεύσει τις ε, ομάδα εργασία για τον ανταγωνισμό. Ο στόχο μα είναι να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε συμφωνία στα πλαίσια των διαδικασιών ε, ε, των κανονισμών εξουσιοδότησης και διαδικασίες και οι δύο σχετικές προτάσεις σε σχέση με αυτούς τους κανονισμούς εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 5 Δεκεμβρίου. Πρέπει να σας πω ότι δεν ακολούθησαν αυτή την πράτη ήθη νομοθετική διαδικασία, αλλά μπορώ να σας εξασφαλίσω ότι η, η πρόθεσή μας είναι να ακούσουμε τα σχόλιά σας και τις ανησυχίες σας. Αυτό σημαίνει πόση σημασία προσδίδει η Ιρλανδία στην ε, δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων και κλίματος στην Ευρώπη για να προωθήσουμε την ανάπτυξη και την θέση απασχόληση. Θα ήθελα σας ευχαριστήσω που με ακούσατε και δίνω αμέσω το λόγο στον συνάδελφο Σεν Σέρλοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετισμό σε κελτική γλώσσα. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας για την πρόσκληση που μας απίφθηνε να, σας, ε, να προσέλθουμε σήμερα εδώ. Και είναι ιδιαίτερη ευχαρίστηση που έχω την τιμή να απευθύνω τον λόγο σε εσά για τις προτεραιότητες για την έρευνα και το διάστημα. Είχα ήδη πέρσι τη δυνατότητα να συναντηθώ με την κυρία Σαρτόρη, επικεφαλής της Επιτροπής σας, καθώς και τους συγητάς Έλερ και Καρβάλιο, και επίσης είχα την ευκαιρία σήμερα το πρωί να συναντηθώ άλλους εισηγητές όπως τον κύριο Ρέμεκ, την κυρία Μαντουρέλ, Ματίας, τον κύριο Σκίνερ. Επίσης, αντιπροσωπεία της Επιτροπής σας ήρθε στο Δουβλίνο τον προηγούμενο Οκτώβριο. Όλες αυτές οι συναντήσεις απαιτέλεσαν την βάση για μια συνεννόηση για κοινούς στόχους. Τώρα για τις προτεραιότητες για το διάστημα. Ως υπουργό αρμόδιος ε, για τα θέματα αυτά, θα ηγηθώ των εργασιών του Συμβουλίου. Η στόχη της Ιρλανδικής Προεδρίας για την πολιτική του διαστήματος είναι να προωθηθεί η σχετική νομοθεσία, να εξασφαλιστεί ε, η απάντηση στο ερώτημα εάν το θέμα θα ενταχθεί στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ή όχι. Και αναμένουμε ότι η Κομισιόν θα υποβάλει σχετική πρόταση μέχρι την άνοιξη του 2014, καθώς επίσης και για την εποπτεία και παρακολούθηση του, στο διάστημα, σημαντική για τους δορυφόρους, την βιομηχανία αλλά και για το κοινό. Επίσης, να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την βιομηχανική πολιτική του διαστήματος, κρίσιμη συνιστόσα που θα βοηθήσει να αυξηθεί η δραστηριότητα των μικρών και μεσών επιχειρήσεων στον τομέα του διαστήματο. Στη διάρκεια τη Προεδρία μα έχουμε τη φιλοδοξία να συμφωνήσουμε επί συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΕΣΑ, που θα προσφέρει προσανατολισμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια σειρά δράσεων που θα επιτρέψει την συνοχή και συμπληρωματικότητα μεταξύ των εργασιών των δύο αυτών οργανισμών και ελπίζω ότι θα μπορέσει να τεθεί αυτό υπόψη των Υπουργών Ανταγωνισμού τον Φεβρουάριο και τον Μάιο. Σημαντική πρόοδος στα ντουσία αυτά θα σημαίνει για μας σημαντική πρόοδο για, την, ε, για το διάστημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν θα πρέπει να λησμονούνται ούτε να υποτιμώνται εδώ οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Στη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας θα συνεχίσω να παρακολουθώ την ανάπτυξη του ε, τομέα του διαστήματος και τα σημαντικά ωφέλη που θα προσφέρει αυτή η ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, στον τομέα της έρευνας και στην κοινωνία και βραχυπρόθεσμα αλλά και πλέον μακροπρόθεσμα. Για τις προτεραιότητες έρευνας και καινοτομίας που αυτά είναι μεγάλη σημασία λόγω του ρόλου που παίζουν στην οικονομική ανάκαμψη, ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιρλανδική Προεδρία έχει τον στόχο εδώ Πρώτα να επιταχύνει την υλοποίηση της δημιουργίας αξίας οικονομικής και κοινωνικής. Δεύτερο, να αυξήσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, να ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και να μεγιστοποιήσει τις συνέργειες μεταξύ των επιπέδων ε, κοινωτικού, εθνικού κλπ. Για να επιτύχουμε στους στόχους αυτούς θα δώσουμε προτεραιότητα στις εξής δράσεις μέσω νομοθετικού έργου, συζητήσεων πολιτικής και συμπερασμάτων του Συμβουλίου και βεβαίως και με συγκεκριμένε ε, εκδηλώσεις για τον ορίζοντα 2021 για την πρόοδο και ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, για ε, σημαντικές enabling technologies όπως νανοτεχνολογία καθώς και η διάθεσή τους στην εμπορία, προώθηση της δυνατότητας καινοτομιών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ενίσχυση της ε, δραστηριότητας των ευρωπαϊκών περιφερειών με μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας. Για τον ορίζοντα 2020 τώρα, βεβαίως, η κέρια προτεραιότητα εδώ για την Ιρλανδική Προεδρία θα είναι να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία για την δέσμη μέτρων για τον ορίζοντα 2020. Ήδη μεγάλο έργο έχει επιτελεστεί από τις προηγούμενες προεδρίες για να υπάρξει κοινή θέση του Συμβουλίου για τα διάφορα τμήματα των ε, προτάσεων για τον ορίζοντα 2020. Η Ιρλανδική Προεδρία θα συνεργαστεί με τις χώρες μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να υπάρξει συμφωνία μέχρι τέλους της Προεδρίας μας για όλο το φάσμα μέτρων του ορίζοντα 2020. Η επίτευξη συμφωνίας για το θέμα αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Έρευνα και κοινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τον ορίζοντα 2020 για να υπάρξει ανάπτυξη με τις σημαντικές flagship πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Είναι προς το συμφέρον όλων μας να μεγιστοποιήσουμε τη χρηματοδότηση για έρευνα και ανάπτυξη. Ιδιαίτερα με ικανοποίησε το γεγονός ότι η Επιτροπή Ήτρε όταν ενέκρινε τη διαπραγματευτική της εντολή τον Νοέμβριο για τον ορίζοντα 2020, έδωσε μεγάλη υποστήριξη στον ορίζοντα 2020 και παραθέτω από αυτά που είπατε, το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ευκαιρία για την Ευρώπη να επενδύσει στο μέλλον της και να της επιτρέψει να εξέλθει από την κρίση. Η πολιτική θα πρέπει να απηχεί αυτόν τον φιλόδοξο στόχο. Γνωρίζω ότι οι συζητήσεις στου τριμερεί διαλόγου έχουν αρχίσει στο τεχνικό επίπεδο για τον ορίζοντα 2020 και η πρώτη προβλέπεται στι 31 πρώτου φέτο Είναι κοινή η δεσμευσή μα για να προωθήσουμε τι διαπραγματεύσει αυτέ και είναι σημαντικό να δείξουμε στους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι εκπροσωπούμε τα δικά του συμφέροντα με τρόπο επαρκή και αποτελεσματικό. Είναι επίση σημαντικό να επιτύχουμε πρόοδο το δυνατόν ταχύτερο έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει επαρκής χρόνος για να προωθηθεί και η απαραίτητη νομοθετική διαδικασία για να αρχίσει η εφαρμογή των σχεδίων αυτών από τις αρχές του 2014. Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με πολλά από τα στοιχεία της προτάσεως πλαισίου, τα ακούσαμε αυτά στο Συμβούλιο, η Ελλανδική Προεδρία αναμένει καρποφόρο συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό το μεγάλο ντοσχέ, και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εξασφαλίσουμε ώστε η εργασία επί των διαφόρων συνιστοσών του πακέτου να συνεχίσει με τις τρεις προτεραιότητε προτεραιότητες του ορίζοντα 2020. Μαζί πρέπει να ενισχύσουμε την υπεροχή της ε, Ευρωπαϊκής Βάσης Έρευνας, την πρωτοπορία στο βιομηχανικό τομέα, και να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες κοινωνιολογικές προκλήσεις με νέες καινοτόμες λύσεις που θα επιτρέψουν ταχύτερη ανάπτυξη και δημιουργία απασχόλησης. Τονίζουν προκειμένου τη σημασία της αρχής της απλοποίησης ως προτεραιότητας. Είναι σημαντικό να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ απλοποίησης και ευελιξίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την επιτυχία του ορίζοντα 2020. Τώρα για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Χρειάζεται τον χώρο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει τα ταλέντα και την επένδυση και τις επενδύσεις για να δημιουργηθεί μια πραγματική ενιαία αγορά γνώσης, έρευνας και καινοτομίας. Η Προεδρία μας γι' αυτό περιλαμβάνει και την παραπέρα εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας μεταξύ των προτεραιοτήτων της, έτσι ώστε να επιτύχουμε σημαντική πρόοδο για την επίτευξη των στόχων που έχει θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήδη από το 2011. Από το 2014 και μετά να αρχίσουν να λειτουργούν τα σχέδια αυτά για να δημιουργηθεί αυτή η ενιαία αγορά γνώσης και καινοτομίας. Καθώς και για τους σχετικούς στόχους της ERA. Έχουμε και άλλες ανοιχτές προκλήσεις όπως την ανοιχτή αγορά για τους ερευνητές και την ενίσχυση της εθνικής συνεργασίας. Προτείνουμε να διεξαγάγουμε συναντήσεις το Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας στις 18 και 19 Φεβρουαρίου και στις 29 και 30 Μαΐου. Θέματα στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας θα είναι καλύτερη πρόσβαση στην επιστημονική γνώση, συζητήσεις θα γίνουν στο Συμβούλιο για το μέγα αυτό θέμα. Η Προεδρία θα συνεχίσει να ανταλλάσσει απόψεις με την Ευρωβουλή έτσι ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω πολιτική για τη λεγόμενη open access και την εφαρμογή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 για να εξασφαλίσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο συντονισμένες δημόσιες επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη. Θα διεξαγάγουμε μεγάλη συνδιάσκεψη από 2 Φεβρουαρίου μέχρι 1 Μαρτίου για τα διδάγματα του παρελθόντος αλλά και την πορεία προς τα εμπρός. Προτείνουμε συζήτηση περί πολιτικής στο Συμβούλιο τον Μάιο. Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική φύση των επενδύσεων για την καινοτομία στην Ευρώπη, η Προεδρία θα προτείνει συμπεράσματα του Συμβουλίου για την στρατηγική φύση του High Performance Recruiting για την καινοτομία, δηλαδή ε, εξέβρεση ερευνητών. Επίσης, είναι σημαντικά τα θέματα αυτά και διευρωπαϊκά. Παίζουν σημαντικό ρόλο για την εξασφάλιση ποιότητας της ευρωπαϊκής έρευνας, καθώς επίσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Η Προεδρία μας θα προτείνει συμπεράσματα του Συμβουλίου για να ενισχύσει τη στρατηγική αυτή για την επίτευξη διεθνών συνεργασιών όπως έχει πει και η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της ERA και να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη διεθνή συνεργασία στην έρευνα και καινοτομία. Εν συμπεράσματι, θα διεξαγάγουμε και άτυπο συμβούλιο για την ανταγωνιστικότητα στις 2 και 3 Μαΐου στο Δουβλίνο, ευθυγραμμισμένα με τα θέματα γενικά της ελληνικής Προεδρίας. Το θέμα του Συμβουλίου αυτού θα είναι πώς να βελτιστοποιηθούν τα ωφέλη από τις ευρωπαϊκές επενδύσεις για να υπάρξει ανάπτυξη οικονομική και κοινωνική. Ελπίζω πολύ η πρόεδρος σας, η κυρία Σαρτόρη, να έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε αυτές τις εργασίες. Ευχαριστώ τον Υπουργό Ρίτσαρτ Μπράτον και τον Υπουργό Σον Σέρλοκ και φυσικά οι ευχαριστίες αφορούν όχι μόνο εμένα προσωπικά αλλά και το σύνολο της Επιτροπής μας. Ο συνάδελφος Ρούμπικ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις δηλώσεις σας. Η Ευρώπη που βρίσκεται τώρα σε κρίση χρέους και ανεργίας έχει ανάγκη από μια ικανή προεδρία. Να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ξανακάνουμε, να ενισχύσουμε τους ανέργους, να μπορέσουν να ξαναγίνουν ανεξάρτητοι, να φροντίσουμε για την επιβίωση των επιχειρήσεων. Η Κομισιόν έχει υποβάλει έκθεση για την, για τον, για την εκ νέου εκβιομηχάνηση της Ευρώπης που είναι σημαντική. Με ενδιαφέρει λοιπόν ποια είναι η θέση της ε, ε, Ιρλανδική Προεδρία για την έκθεση COSME όπου το Κοινοβούλιο έχει γράψει 4 δισεκατομμύρια και η Κομισιόν προβλέπει το μισό από το ποσό αυτό. Επίσης, τι πιστεύετε για την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για διάθεση 100 δισεκατομμυρίων για τον ορίζοντα 2020 αντί των 80 που προβλέπονται τώρα. Θα με ενδιαφέρει επίση να μάθω το πρόγραμμα Έρασμο για νεώρου επιχειρηματίες. Δεν μπορεί να θεωρηθεί και αυτό προτεραιότητα. Θα μπορέσει να δώσει με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα σε νέους να πάνε σε άλλες χώρες να διδαχτούν πώς γίνεται κανείς επιτυχημένος επιχειρηματίας. Διότι δυστυχώς η Ευρώπη πάσχει από έλλειψη επιχειρηματιών και υπερπληθώρα ανέργων. Αυτό που μας χρειάζεται είναι απασχόληση. Με ενδιαφέρει λοιπόν με ποιον, με τι προετοιμάζει η Προεδρία σας ε, στα θέματα αυτά. Ähm, Ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα προσεκτικά και χαίρομαι που είπατε ότι θέλετε να προχωρήσετε στον τριμερή διάλογο για τον ορίζοντα 2020 και τα σχετικά προγράμματα. Πράγματι υπάρχουν πολλά κολλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν. Θα βοηθήσει πολύ εάν μέσα στα πλαίσια της Προεδρίας σας ασχοληθείτε εντατικά για να διαμορφώσετε πλειοψηφίες και για τη χρηματοδότηση. Για τη στρατηγική του διαστήματος και γενικά για τα μεγάλα έργα. Έχουμε τρία έργα που πρέπει να συζητήσουμε την μελλοντική τους χρηματοδότηση και από πού θα προέλθει αυτή. Πρόγραμμα Γαλιλαίος, επίσης Global Earth Monitoring System, καθώς και το ITER. Ακούγονται διάφορες παραλλαγές εντός ή εκτός του κοινοτικού προϋπολογισμού. Για το EGMS έχουμε ζητήσει ως Κοινοβούλιο να μπει μέσα στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ερωτώ ποια θα είναι η θέση σας. Θα ταχθείτε μαζικά υπέρ αυτής της ιδέας, θα αναζητήσετε κάποιες πλειοψηφίες είτε προς τη μια είτε προς την άλλη κατεύθυνση στο Συμβούλιο. Και το τρίτο, για το EAGMS, να ασκήσετε κάποια επιρροή στην Κομισιόν και στον Πρόεδρό της για να καταθέσει το σχέδιο κανονισμού για τον οργανισμό αυτό. Διότι κάποια στιγμή πρέπει να συζητηθεί. Φαίνεται πως ήδη έχει προχωρήσει αρκετά. έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για την παρουσίαση των προτεραιτήτων της ε, Ιρλανδικής Προεδρίας. Νομίζω πως όλοι εμείς ε, στο Κοινοβούλιο δεν μπορούμε παρά να υποστηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα το τόσο φιλόδοξο της Προεδρίας. Έχω κάποια σχόλια σχετικά με τον ορίζοντα 2020. Πράγματι έχει ιδιαίτερη σημασία να προχωρήσει παράλληλα με την καινοτομία αλλά και με τα νέα startups που συνδέονται με τον ορίζοντα 2020 αλλά και να μπορέσουμε να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία στο πλαίσιο του προπολογισμού και ρωτώ την Προεδρία τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως Κοινοβούλιο, όπως είπε ο κύριος Ρούμπικ, αποκοινούμε την Προεδρία για να υπάρξουν αυτές οι επενδύσεις που είναι τόσο απαραίτητες για την κοινοτομία και την έρευνα. Και μια δεύτερη ερώτηση πάντα στο αυτό πεδίο αναφορικά με την συμμετοχή στην έρευνα δεν θα πρέπει αυτή να γίνεται μόνο σε γεωγραφικό επίπεδο, αλλά υπάρχουν και μικρά Ινστιτούτα, πανεπιστήμια κλπ. Πώ μπορούν να συμμετέχουν αυτοί οι οργανισμοί, αυτά τα ιδρύματα. Είδαμε πως η, η Ιρλανδία έχει αποκτήσει εμπειρία σε ζητήματα καινοτομία και έρευνα. Στο κοινοβούλιο μα ίσως να έχουμε κάπω διαφορετικέ θεωρήσει για το πώς ε, μπορούμε να ασχοληθούμε με τα θέματα της έρευνας. Ίσως και τα διορθωτικά ταμεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ε, για να δοθούν κάποια χρήματα. Και κάτι ακόμα, όταν διατυπώσαμε τους στόχους για τον ορίζοντα 2020, μιλούσαμε για την αύξηση της συμμετοχής από πλευράς βιομηχανιών. Νομίζω ότι παρά την οικονομική κρίση που μαστίζει την ε, Ευρώπη, ε, τονίστηκε το ζήτημα της επένδυσης από πλευράς ε, επιχειρήσεων, ότι βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσης και ρωτώ, θα είναι δυνατόν να προβλεφθούν επενδύσεις από πλευράς ιδιωτών και επιχειρήσεων. Φυσικά η θέση σας έχει ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να πετύχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Λάμπερτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας χαιρετίζω κύριε Υπουργή. Έχω μεγάλες προσδοκίες από την πρόεδρε σας και δεν ήταν πολύ ενθαρρυντική η διάλογοι η τριμερείς. Εχθές έγινε ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Οικονομικών σας και δεν ήταν ενθαρρυντική παρομοίως. Εδώ μιλούμε για μέτρα βελτίωσης της οικονομίας, για την ανάπτυξη, την αναθέρμανση της οικονομίας της Ευρώπης. Θα ήθελα να εστιαστώ στον ορίζοντα 2020. Το πρώτο σχόλιο από τα διαπραγματεύσεις είναι ότι δεν είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί στις 31 του μηνός. Η προεδρία σας, πρέπει να σας πω, ότι χρησιμοποιεί τρεις εβδομάδες για να προετοιμαστεί, αλλά η στάση του Συμβουλίου που εκπροσωπείται είναι ξερέσουμε τα τεχνικά θέματα είναι ότι πιστεύετε ότι δεν είναι καλή ιδέα αυτή. Πραγματικά θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να διαβάσετε αυτά τα οποία γράψατε εσείς. Δεν είμαστε άσχετοι. Μπορεί να έχουμε κάποιες καλές ιδέες και μπορεί να είχαμε έρθει και σε επαφή και να έχουμε και την άποψη κάποιων μελών του Συμβουλίου. Εσείς είπατε ότι δεν έχουμε τέτοιου είδους εξουσιοδότηση διαπραγματεύση, αλλά νομίζω ότι καλύτερα θα είναι να αναθεωρήσετε κάπως πριν αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις την επόμενη εβδομάδα. Σε κάτι άλλο να εστιάσουμε, στις ΜΜΕ. Όλοι οι πολιτικοί λέγουν ότι η ΜΜΕ είναι πολύ έτσι χρειαζόμαστε, εδώ εκφράζεται η καινοτομία, είναι στον πυρήνα της οικονομίας. Αλλά την ώρα της αλήθειας βλέπουμε ότι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ε, χάρη στις δυνατότητες λόμπι που έχουν κάνουν τα πράγματα να γυρίσουν προς όφελός τους. Ελπίζω λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύτων ορίζοντα 2020 το Συμβούλιο θα έρθει να μας ε, συναντήσει όχι στο τέλος διαδικασίας αλλά θα συμφωνήσει με αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε. Να τους δώσουμε καλή χρηματοδότηση, περισσότερο από τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να βοηθηθούν διαφορετικά και όχι μόνο με κονδύλια. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε αυτό να το επιτύχουμε και τελειώνοντας θα πω το εξή. Πιστεύω ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να είναι σύμμαχοι. Τι διαπιστώνετε και αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται σε επίπεδο όλων των θεσμικών οργάνων. Πολλές φορές ανταλλάσσουμε απόψεις για να δούμε ποιος θα πάρει ποιο κομμάτι και ποιος είναι υπεύθυνο για κάθε κομματιόν. Σε επίπεδο όμως των ΜΜΕ αποδείχθηκε ότι το καλύτερο όπλο που έχει η Επιτροπή για να προχωρήσει σωστά είναι να μιλάει σωστά με τις ΜΜΕ. Και στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 δεν θα ήθελα να αναθέσει ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα και τις ΜΜΕ η Επιτροπή σε κάποιον άλλο οργανισμό. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα μέσο το οποίο έχουμε, το οποίο είναι σωστό, δουλεύει και να μην αρχίζουμε να λέμε κάτι διαφορετικά, διαφορετικό. Ελπίζω ότι μπορώ να υπολογίζω στη δική σας υποστήριξη και να είναι ενδιαφέροντα αυτά που θα κάνουμε το παρόν εξάμεινο. Ευχαριστώ. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη με την ένταξη της Ιρλανδικής Προεδρίας. Αυτή είναι μια μέρα την οποία πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα φιλόδοξοι. Είμαι πάρα πολύ φιλόδοξη για τον ορίζοντα 2020. Διάβασα αυτό το βιβλίο το οποίο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και αυτό είναι το τελευταίο αντίτυπο. Μπορώ να σας το προσφέρω. Αφορά το ζήτημα της έρευνας, τεχνολογίας και της, της και της χρηματοδότησης. Χαίρομαι που το Ευρωκοινοβούλιο ζήτησε κάποιες ε, μετακινήσει σε κονδύλια στον προπολογισμό. Όπως ε, είπε και ο Υπουργό σήμερα το πρωί, ένα από τα ζητήματα που μας απασχολεί είναι το θέμα το ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να εμπίπτουν πάντα στις οδηγίες και να εξαιρούνται από κάποιες από αυτές. Συχνά λέμε ότι θέλουμε να τις απαλλάξουμε. Υπουργέ. Αλλά θα πρέπει τελικά να βρούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες και να δούμε ποιες ε, μικρές θα πρέπει να απαλλαχθούν και βέβαια καταλαβαίνετε και γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτή είναι μια συζήτηση ιδιαίτερα περίπλοκη. Παρακαλώ λοιπόν στο πλαίσιο αυτή τη θετική, θετικού οράματο περί ανταγωνιστικότητας βοηθήστε μας ε, να ε, προωθήσουμε κάποιες εξαιρέσεις ε, και για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. κυρία Καρβάγιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργοί, συνάδελφοι, αρχίζοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την παρουσία τους στους Υπουργούς και διότι μας εξηγούν τις προτεραιότητες τις Προεδρίες γιατί αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα για την Ευρώπη. Είμαι η συγγήτρη για το πρόγραμμα Horizon 2020 και προσβλέπω σε επιτυχείς διαπραγματεύσεις και ελπίζω πραγματικά ότι θα είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε το πακέτο αυτό κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ καρποφόρα συνεργασία που είχαμε στα πλαίσια προετοιμασίας της Προεδρίας σας και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα. Όπως ίσως γνωρίζετε, υπάρχουν θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την πολιτική μας ομάδα. Ήδη το ένα το ανέφεραν οι συνάδελφοι, η ειδική συμμετοχή βιομηχανία των ΜΜΕ έχουμε το κατάλληλο μέσο που μας το επιτρέπει αυτό και απλούστεροι μηχανισμοί για τις ΜΜΕ. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα είμαστε σε θέση να έχουμε για τις ΜΜΕ ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα και θα μπορέσουμε να τη συμπεριλάβουμε σε όλες τις φάσεις του προγράμματος. Το δεύτερο θέμα αφορά την ε, ε, αριστεία και το πώς μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση. Χαιρετίζουμε την οποιαδήποτε πρωτοβουλία χωρίς άλλες ε, εκ των προτέρων προϋποθέσεις. Είναι πρωταρχική σημασία να ενθαρρύνουμε όσους πάρουν τα βραβεία αριστείας να συμμετάσχουν στις πρωτοβουλίες, γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί να τις βοηθήσει τις επιχειρήσεις αυτές να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Horizon 2020. Και γι' αυτό έχουμε συμπεριλάβει μέτρα που θα διευκολύνουν την νέους να έχουν πρόσβαση και τους τρόπους με τον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω αδελφοποιήσεων κτλ. κτλ. Έχουμε πάρα πολύ φιλόδεξη προγράμματα καλύπτοντας όλο τον τομέα των καινοτομιών και προγράμματα τα οποία όχι μόνο στα πλαίσια του, ορίζ, του προγράμματος Horizon 2020 θα πρέπει να κινητοποιήσουμε με κοινή συμμετοχή και με συγχρηματοδότηση καθώς και σχέδια και προγράμματα επίδειξης με τη δημιουργία συνεργειών ώστε εάν κάποιες επιχειρήσεις θέλουν να συγχρηματοδοτήσουν προγράμματα να μπορούν να το κάνουν στα πλαίσια ενός προγράμματος, στα πλαίσια πιο απλοποιημένων διαδικασιών, γιατί όλα αυτά ήταν πάρα πολύ πολύπλοκα. Έχουμε τους σχετικούς κανονισμούς και στα πλαίσια του γράμματος ορίζων 2020 και των περιφερειακών ταμείων θα πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιούμε με απλούστερο τρόπο τους πόρους που χρειάζονται. Μιλήσατε για απλοποίηση. Εγώ ήμουν επίσης εισηγήτρια για την απλοποίηση. Θέλουμε η απλοποίηση για τους χρήστες να έχει τις σωστές προτεραιότητες, να είναι απλή, σωστά δομημένη σε όλους τους τομείς, την απλή, στην εφαρμοσμένη έρευνα, κυρίως στα πλαίσια του προγράμματος Ορίζον 2020. Επίσης, χρειαζόμαστε τα κατάλληλα κονδύλια για να ολοκληρώσουμε όλες αυτά τα σχέδια που έχουμε και υπολογίζουμε σε εσά για να μας συνδράμετε. Ξέρω ότι εσείς προσδίδετε ως χώρα μεγάλη σημασία στην έρευνα. Γι' αυτό να μας βοηθήσετε για να αποφασίσουμε το μέλλον της έρευνας στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να συγχαρώ τους Ιρλανδούς υπουργούς και να τους καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Ξέρω ότι αυτή η περίοδος που διανύουμε είναι δύσκολη αλλά και συνάμα πολύ σημαντική. Συζητήσαμε θέματα τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουν βρει τη λύση τους και δεν νομίζω ότι θα κατορθώσετε να τα επιλύσετε καρδιά και δική της προεδρίας. Τώρα σκεπτόμενοι το μέλλον ίσως ε, να κανονίσουμε, να επιταχύνουμε την επίλυση κάποιων ε, προβλημάτων τώρα για τον ορίζοντα 2020 ε, και το σχετικό πρόγραμμα. Δεδομένη τη δύσκολη οικονομική κατάσταση και τη ύφεση που επικρατεί, οι διαπραγματεύσει θα είναι περίπλοκε. Αλλά το πρόγραμμα θα διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον προκειμένου να βοηθήσει τις οικονομίες μας να ανακάμψουν. Και οι προσπάθειές σας προκειμένου να υπάρξει συντονισμός όλων των δράσεων είναι, όπως καταλαβαίνετε, ιδιαίτερα σημαντικό. Δεν έχουμε ακόμα χρησιμοποιήσει πλήρως το, τις δυνατότητες αυτού του προγράμματος. Συνεχίζουμε να χάνουμε ε, αντιγνωστικότητα απέναντι σε άλλες χώρες ε, και ειδικά σε, αναδυνο, σε οι οποίες χρηματοδοτούν την ε, ακαδημαϊκή έρευνα με τρόπο πιο αποτελεσματικό. Εάν δεν επενδύσουμε λοιπόν, τότε θα περάσουμε στην περιφέρεια αυτού του κλάδου. Η Ευρώπη της έρευνας. Η Ευρώπη δεν η δεν είναι πια ελκυστικός πόλος ε, για ακαδημαϊκούς ε, που ασχολούνται με έρευνα. Ε, οι μισθοί, παραδείγματος χάρη, είναι χαμηλότεροι σε πολλές περιπτώσεις. Ε, δεν υπάρχει κίνητρο για τους επιστήμονες να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λείπει η πολιτική βούληση και δεν λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των αγορών μας. Να σας ρωτήσω τώρα για το ποια θα είναι, ποια είναι η για τα πράγματα που αφορούν στον ορίζοντα 2020 και τι γνώμη έχετε για τις αρχές που θα πρέπει να αποτελέσουν την βάση για την μελλοντική ευρω... Ε, στρατηγική έρευνας και να καταστούμε πόλος έλξης ε, της επιστημονικής κοινότητας. Πρέπει να εξετάσουμε και τα πλεονεκτήματα των προγραμμάτων που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από μας. Παρακαλώ. Ο κύριος Έλερ. Ευχαριστώ στα αγγλικά. Σας ευχαριστώ για την προσέλευσή σας εδώ. Στο Κοινοβούλιο είχαμε την εντύπωση στα πλαίσια της προετοιμασίας της Ιρλανδικής Προεδρίας ότι τα πήγατε πολύ καλά. Και αναμένουμε με, ιδιαίτερα, με, ιδιαίτερη, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σας δούμε να δουλεύετε ε, ε, πραγματικά με αυτή την ε, ευελιξία και, την, και το ρεαλισμό που σας διακρίνει. Τώρα έχω δύο βασικά θέματα για την πρόταση ορίζοντας 2020. Πρώτα, κατανοείτε ότι κατά κάποιο τρόπο ορίζοντας 2020 είναι μοναδικός, γιατί δεν είναι αυτό το γενικό. Ακόμα και τα προγράμματα CIP και τα λοιπά, έχουμε να βάλουμε συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις. Θα γνωρίζετε επίσης ότι, ότι αυτά τα δεδομένα καλάθια για το διαπραγματεύσεων και τα δεδομένα νούμερα της, των, του Συμβουλίου είναι τρομερά θα έχουν τρομερές επιπτώσεις. Δεν αναμένω να σχολιάσετε αυτά τα πράγματα τώρα βέβαια ιδιαίτερα εντατικά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η διάσταση περικοπών που προτείνονται τώρα δεν οδηγούν σε μια αντιμετώπιση του Κοινοβουλίου που να δέχεται οριζόντιες περικοπές. Δεν μπορείτε να αναμένετε ότι θα τα δεχτούμε, θα κάνουμε αναλογικές περικοπές και θα καταλήξουμε με υποχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Τι αναμένεται λοιπόν ως έκβαση του πολίτους δημοσιονομικού πλαισίου γύρω στα 70 δισεκατομμύρια και λιγότερα. Έχετε για παράδειγμα υπόψη στην επιλογή ε, να βγάλετε την κοινή αγροτική πολιτική έξω ε, επίσης το GMS ή άλλα πράγματα όπως πρότεινε η Κομισιόν ποιες είναι οι προσδοκίες σας, εάν δηλαδή έρθουμε να συζητήσουμε τις περικοπές, με ποιο τρόπο θα τις, θα, τις ε, υλοποιήσουμε. Επίσης υπάρχουν υψηλές προσδοκίες για την Ιρλανδική Προεδρία, παρόλο που γνωρίζουμε ότι γνωρίζετε τα προβλήματα που προκαλούν οι πολιτικές λιτότητες και τα σοβαρά προβλήματα των ε, δημόσιων προπολογισμών. Παρ' όλα αυτά, εάν καταλήξετε τελικά στα νούμερα που προτείνει το Συμβούλιο, γνωρίζω θα φτάσουμε και κάτω από το 1,8% του ΑΕΠ. Είμαστε λοιπόν ακόμα πολύ μακριά από αυτά τα 3%. Η αντίδραση δεν είναι απλά αντίδραση πάνω στον προϋπολογισμό, θα είναι άμεση αντίδραση και των αγορών. Διότι θα αναρωτηθούν κατά πόσο ο προϋπολογισμός αυτός έχει κάποια σχέση με ανάπτυξη και θα αρχίσει μια ευρύτερη συζήτηση για την σχέση μεταξύ ανάπτυξης, ανάπτυξης και του ορίζοντα 2020 και του πυλώνα 1. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη λέει ναι, καινοτομία κτλ. Ωραία λόγια. Αλλά στην πράξη υπάρχει μια πτυχή ανάπτυξης. Αν μείνουν όλα σε τομείς όπως η κοινή αγροτική πολιτική κτλ. δεν θα υπάρξει ανάπτυξη. Τρίτο, για την απλοποίηση. Είπατε κάπως διπλωματικά, απλοποίηση και ευελιξία. Η θέση του Κοινοβουλίου πάντοτε ήταν υπέρ της απλοποίησης. Η ιδέα που ρίχτηκε αρχικά από το Κοινοβουλίο με την έκθεση Καρβάλιο και μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι ναι μεν θέλουμε την απλοποίηση, αλλά θέλουμε και το ε, λεγόμενο leverage, τη μόχλευση. Αν δείτε τους τελευταίους συμβασμούς του Συμβουλίου που αυξάνεται από 22% σε 25% το άμεσο κόστος και μιλείτε και για έξτρα χρήματα, για μισθολογικά κτλ. και τα μεταφέρει αυτά σε συγκεκριμένα ποσά η Κομισιόν, πάει να πει ότι είναι αυτά 70% του προπολογισμού, 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ρεαλιστικό να αυξάνονται τα έμεσα κόστη σε ένα βαθμό όπου θα έχουμε τελικά λιγότερα κονδύλια για λιγότερα προγράμματα. Και τέλος, παραθέτω κάτι που είπατε. για το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Είπατε για, το, για την ψηφοφορία του 2012 υπό Ολλανδική Προεδρία Είπατε ότι τα πανεπιστήμια εργάζονται για, να, για μελέτες για το κόστος. Ίσως ορισμένα μοντέλα να λειτουργούν για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όμως δεν θα λειτουργήσει για μεγάλες επιχειρήσεις και θα αποτελέσει αποτροπή για τη συμμετοχή τους στην ορίζοντα 2020. Άρα η θέση του Κοινοβουλίου τελικώ απηχεί την θέση τη Ιρλανδική Προεδρία. Ε, Ευχαριστώ. Ο κύριο Σέντο Ιαλαμπάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα σχόλιο να κάνω, διότι πολλές από τις ερωτήσεις ε, που προέβλεπα να κάνω ε, αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους σου σχετικά με τον προϋπολογισμό. Εμείς δάμε να αυξηθεί φυσικά ο προϋπολογισμός για το 2020. Θα ήθελα να υπογραμμίσω πως αν θέλουμε η έρευνα να έχει μια σωστή αντιμετώπιση, σημασία έχουν και οι εθνικοί προπολογισμοί στον τομέα της έρευνας. Προέρχεται από μια χώρα όπου γίνονται ικανοποιητικέ δαπάνε στον τομέα τη έρευνα, αλλά σε περίπτωση, μάλλον στην περίπτωση αυτή, λόγω τη οικονομική κρίση, είναι δύσκολα να διατηρήσουμε τους εθνικούς αλλά και τους περιφερειακούς προπολογισμού σε ικανό επίπεδο. Μπορεί να κάνουμε προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά χρειάζεται να διατηρήσουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο επενδύσεων και σε εθνικό και στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Τόγια, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου προς την ε, Ιρλανδική Προεδρία. Είχαμε την ευκαιρία να τη συναντήσουμε και να συζητήσουμε τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και σε άλλους χώρους. Δύο παρατηρήσεις. Ε, μια παρατήρηση και ένα αίτημα. πρώτη παρατήρηση αφορά, όπως είπαν και πολλοί συνάδελφοι, το, το θέμα του προπολογισμού για τα κεφάλαια και τα προγράμματα τα οποία ε, μπορούν να δώσουν κάποια όθηση στον τομέα της ανταγωνιστικότητα και τη ε, απασχόλησης. Ε, για να είμαστε και συνεπείς στο κάτω-κάτω δεν υπάρχει έγγραφο, ομιλία, πρόγραμμα που να μιλάει για αύξηση της απασχόλησης, αλλά έχουμε αυτό το πρόβλημα του προπορισμού για το ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που είναι κάπως σχιζοφρενικό. Ε, ξεκινήσαμε από τα αιτήματα του Κοινοβουλίου, της προτάσεις Κομισιόν για τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές, μια πρόταση σχετικά με το ορίζοντα 2020, αλλά τα πράγματα πηγαίνουν όπως προβλέπαμε. Τα κράτη-μέλη κινητοποιούνται προκειμένου να στηρίξουν μια ανανεωμένη ΚΑΠ, το στόχο της συνοχής και το ορίζον 2020 παραμένει δίχως ε, πατρότητα. Θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι αυτή η πατρότητα, η μητρότητα, όπως θέλετε. Τώρα, το δεύτερο θέμα αφορά κάπως την πρακτική. Όπως είπαν κάποιοι συνάδελφοι, ε, τόνισαν τα ισχυρά σημεία του προγράμματος Ορίζοντα 2020 και μία ερώτηση συγκεκριμένη. Επειδή έγινε σωστή επιλογή και η συμπληρωματικότητα της μικρόψης επιχειρήσης για την κοινοτομία αφενός του πρόγραμματος ορίζοντα 2020 και του κόσμου, αλλά και για τα διαφορετικά ταμεία, πρέπει να είμαστε σαφείς επί του Δήμαρχου, διότι η συμπληρωματικότητα είναι πολύ ωραίο πράγμα, χρήσιμο. Αλλά <clears throat> αν δεν χρησιμοποιηθεί με τρόπο σωστό και αποτελεσματικό, τότε υπάρχει δυνατότητα σπατάλης πόρων. Να δοθούν λίγα από εδώ, λίγο από εκεί και στο τέλο να μην βρεθούν τα κατάλληλα κονδύλια για την ε, συνεργασία των δύο αυτοκλάδων. Θα πρέπει λοιπόν να έχω κάποιε πιο σαφεί ιδέε από πλευρά σα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, για την καινοτομία ιδιαίτερα στο πλαίσιο του Horizon και την δυνατότητα χρησιμοποίηση των διαθωτικών πόρων συμπληρωματικά. Εν περιπτώσει κάποια στοιχεία διαφάνειας ε, θα πρέπει να μας παρέχεται ω Προεδρία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλλη έχει το λόγο. Ο κύριος Κέλλη ομιλεί την Κελτική. I'm not sure uh, Νομίζω ότι δεν υπάρχει διερμηνία από τα κελτικά, παρατηρεί ο κύριος Κέλλη. Έχουμε δύο υπουργούς, τους καλωσορίζω. είναι αποτελεσματικότατη υπουργή, θα το καταλάβατε από τις παρουσιάσεις τους τώρα προς τον κύριο Μπράτον να πω ότι είναι πολύ σωστό να μειωθεί το άχθος προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά εμείς με αυτά που κάνουμε είναι να δημιουργούμε περιττέρω άχθος με την νομοθεσία που στηρίζουμε τον τελευταίο καιρό και από τις μελέτες αντικτύπου και από τις συναντήσεις που είχαμε σήμερα το πρωί διαπιστώσαμε ότι αν θέλουμε να εφαρμόσουμε τις προτάσεις αυτές θα οδηγηθούμε σε ένα μεγαλύτερο διοικητικό άχθος προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία εδώ και καιρό διδάσκουμε και στην περίπτωση αυτή φυσικά θα έχετε την πλήρη στήριξη της Επιτροπής μας. Ε, τώρα σε όλη τη φορά του κύριο Σέρλοκ αναφερθήκατε στις μικρές επιχειρήσεις ε, και εμείς στην ε, εκλογική περιφέρεια έχουμε μεγάλη εμπειρία περί αυτών Επίσης, ε, ό,τι αφορά το διάστημα, ξέρουμε ότι χρησιμοποιούνται πολλοί οι διάφοροι δορυφόροι και από τους οποίους ε, μπορούν να κερδίσουν πολλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στις συναλλαγές τους τώρα για τον ορίζοντα 2020 θα πρέπει να έχουμε έναν στόχο του 30% για του ΑΕΠ Αλλά παράλληλα έχουμε ακούσει ε, κάποιες φήμες για μείωση των επενδύσεων στον τομέα αυτό. Η διέρευνα, μην ξεχάμε, ότι αφορά όλους τους τομείς, όλους τους κλάδους. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό επιχείρημα όταν θα πρέπει να ε, προωθηθεί και να υλοποιηθεί το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τέλος, προς τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, που μιλούν για συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας και της έρευνας. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Ε, Προτίθεμε να διοργανώσω μια σημαντική διάσκεψη εδώ, στο Κοινοβούλιο, το 4 Μαρτίου, όταν θα έχουμε στη διάθεσή μας το όλο Κοινοβούλιο, θέλετε και ελπίζω με αυτή την προσπάθεια να πετύχουμε μια ευρύτερη συνεργασία ε, υποφελία των πολιτών και για μια καλύτερη χρήση των ε, κονδυλίων που έχουμε στη διάθεσή μας για την επίλυση κάποιων ε, κοινωνιακών ζητημάτων. Και για μια ακόμα φορά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ. άντρε Μπαρέα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ιρλανδική Προεδρία για την ε, παρουσία της. Σήμερα το πήγαμε και κάποιον άλλο συνέλφο. Μία από τις προτεραιότητες πρέπει να είναι η βελτίωση της απασχόλησης, η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, δεδομένου ότι η κατάσταση όσον αφορά την ενεργεία είναι καταστροφική σε πολλές χώρες, κυρίως μεταξύ των νέων που είναι ιδιαίτερα ενισχυτικός. Κατά συνέπεια, τα μέτρα δημιουργίας κινήτρων θα εξαρτηθούν και από τα κονδύλια που είναι απαραίτητα για να δοθούν κίνητρα. Κατά συνέπεια, μία από τις μου είναι ποια συγκεκριμένα μέτρα σκέπτεται να λάβει η Ιρλανδική Προεδρία για να δημιουργήσει τέτοιου κίνητρα. Και βεβαίως, όταν μιλούμε για ανάπτυξη και απασχόληση μιλούμε και για την κινητήρια δύναμη αυτών, της ΜΜΕ. Ποια είναι τα ειδικά μέτρα τα οποία σκέφτεστε να θέσετε σε εφαρμογή για να επαναδροστερηθούν οι ΜΜΕ και να έχουν πρόσβαση στην πιστότηση. Έχετε κάποια συγκεκριμένα μέτρα να προτείνετε, δεδομένου ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Χίμνερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργή, χαίρομαι που ήρθατε στη συνάντηση της Επιτροπής μας και πρέπει να πω ότι ο ρόλος που έχετε αναλάβει στα πλαίσια της Προεδρίας είναι πολύ σημαντικός. Θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε χρόνο και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να βρούμε νέες προοπτικές για τον προπολογισμό. Και έφτασαν και κάποιες φήμες στα αυτιά μας, δηλαδή ότι οι περικοπές θα είναι περικοπές στην εκπαίδευση και στην κοινοτομία. Αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ, διότι πρέπει να σας πω ότι εμείς είμαστε ε, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πλευρά σας και θα υποστηρίξουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία προβλέπεται ώστε να δοθούν χρήματα και να μην περικοπούν αντιθέτω σε θέματα παιδείας και έρευνα. Και θα ήθελα να σας κάνω τις εξής ερωτήσεις τώρα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε πρόταση για να μπορέσουν να επαναδραστηριοποιηθούν τα ερευνητικά κέντρα και κυρίως τα ερευνητικά κέντρα της πρώην Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Διότι ενώ παλιά δεν ήταν σε καλή θέση, αυτή τη στιγμή βλέπω ότι έχουν μεγάλο αποθεματικό εμπειρογνωμόνων και ερευνητών. Δεύτερον, θα θέλαμε στον προπολογισμό να δούμε να έχει την κατάλληλη θέση, τη που τη αρμόζει το πρόγραμμα Horizon 2020. Και θα είναι δύσκολα τα πράγματα αν δεν έχουμε την απαραίτητη υποστήριξη για τις ΜΜΕ. Θα ήθελα να μου πείτε αν η δική σας Προεδρία έχει σκεφτεί τι είδου πρωτοβουλίες πιστεύετε ότι μπορούν να εγκριθούν ώστε όλες αυτές ε, οι καινοτομίε, όλε αυτέ οι νέε ανακαλύψει να μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα, ώστε να μπορέσει να παραμείνει ανταγωνιστική, να εγγυηθούμε την ανταγωνιστικότητα τη Ευρώπη. Διότι εάν γίνει μία νέα ανακάλυψη από κάποιον θα πρέπει γρήγορα εμείς να μπορέσουμε να την διασφαλίσουμε. Δεδομένου ότι ξέρετε ότι υπάρχει πολύ σκληρό ανταγωνισμό από την Κίνα, την Ιαπωνία και τη ΣΥΠΑ. Ευχαριστώ. Τελευταία ομιλητή, η κυρία Χάντεμπορ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα μικρομεσαίε επιχειρήσει ε, για τις οποίες μιλήσαμε σήμερα το πρωί στο γεύμα, στο πρόγευμα μάλλον, εξτάσαμε το ζήτημα της μελέτης αντικτύπου, το οποίο θεωρούν πολλές από αυτές ότι αποτελεί ένα σαφές και στέρεο πλαίσιο Προηγούμενα μίλησα για τον κανονισμό προστασία δεδομένων ΔΙΣ. Δεν θα αναφερθώ περαιτέρω, αλλά ζητάω από την Ιρλανδική Προεδρία να εξετάσει προσεκτικά τι γίνεται με τον κανονισμό περί προστασίας δεδομένων, διότι είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη τις προσδοκίες ε, των πολιτών αλλά και των ψηφοφόρων παράλληλα όμως και των επιχειρήσεων, των εταιριών. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τον γύρο των ερωτήσεων. Υπήρξαν 14 συνάδελφοι που παρενέβησαν. Ε, υποβλήθηκαν πάρα πολλές ερωτήσεις. Ε, έχουμε στη διάθεσή μας τώρα 25 λεπτά για την απάντηση. Well, um... Ευτυχώς, ευτυχώς, οι περισσότερες ερωτήσεις απευθύνονται στον συνάδελφό μου, Σον Σέρλοκ. Θα απαντήσω πάντως σε ορισμένα που μου θέσατε εμένα. Και αρχίζω με τον κύριο Ρούμπιχ, που μίλησε για το μέγεθος του προϋπολογισμού, για τον ορίζοντα 2020. Βέβαια, το μέγεθος του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, της χρηματοδότησής του δηλαδή, θα είναι κρίσιμο για όλα τα, όλες τις χρηματοδοτήσεις που επιθυμούμε να κάνουμε. Συζητήσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο για το μέγεθος του MFF θα επηρεαστούν και από, τις, ε, από τα διαβήματα του Πρόεδρου Βαν Ρόμποϊ αλλά και από τις αποφάσεις του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η ικανότητα που διαθέτουμε δηλαδή στα διάφορα συμβούλια θα είναι κάπως περιορισμένη. Ωστόσο, θα ήταν λάθος να εξετάσουμε μοναχά τα δημοσιονομικά κονδύλια ως πηγή για ανάκαμψη και ανάπτυξη. Το δικό μου χαρτοφυλάκιο, που άπτεται και δύο άλλων συμβουλίων, βλέπουμε δυνατότητες να αναπτυχθεί η ατζέντα του εμπορίου διαπραγματεύσει με τον Καναδά για παράδειγμα που πλησιάζουν στην ε, ολοκληρωσή τους. Επίσης ανοίγουν διαπραγματεύσεις με τις Ενωμένες Πολιτείες και πολλές άλλες χώρες οι οποίες βρίσκονται τώρα σε δυσκολία ατενίζουν τις εξαγωγές ως σημαντική πηγή ε, εσόδων για τις οικονομίες τους. Επίσης, για την ίδια την ενιαία αγορά, η εφαρμογή των διατάξεων της ενιαίας αγοράς και η επέκταση των ρυθμίσεων αυτών, αυτών προσφέρουν επίσης σημαντικές ευκαιρίες στις χώρες μέλη. Και νομίζω ότι πρέπει να εξισορροπούνται και με άλλα μέτρα. Ειδικά για τα προγράμματα των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων, ασφαλώς και υπάρχει, υπάρχει και η ανάγκη ανοίγματο τη πρόσβασης, χρηματοδότηση με σχετικά προγράμματα, αλλά το ίδιο και το πρόγραμμα κοινωνική καινοτομία της επιτροπή Απασχόλησης, των μικροπιστώσεων. Πολλές χώρες αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες πρόσβασης στην χρηματοδότηση από πλευρά των επιχειρήσεών τους. Και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κινείται ωστόσο περισσότερο για να αναπτύξει μηχανισμούς χρηματοδότησης non-bank. Υπάρχει ένας αριθμός δυνατοτήτων που ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να βελτιώσουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και θα αποτελέσει ένα σημαντικό τμήμα της δικής μας ανεπίσημης προσέγγισης, όπως είπα και προηγουμένως, και μετά από συζητήσεις με άλλους η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Τα θέματα των μικρών και μεσών επιχειρήσεων είναι κάτι που δεν πρέπει να μείνει στα λόγια όπως είπε κάποιος από εσά. Πρέπει να αναπτυχθούν συγκεκριμένα μέτρα. Η κυρία Φόρντ και ο Σον Κέλλη έθεσαν το θέμα με την έννοια ότι πρέπει να μειωθεί η επιβάρυνση των μικρών και μεσών επιχειρήσεων. Αλλά βέβαια κάνοντας αυτό ίσως άθελά μας να προκαλούμε άλλες επιβαρύνσεις. Πάντως υπάρχουν, ενθαρρύνομαι από ορισμένε πρωτοβουλίες όπως η Accountancy Directive, η οδηγία για τα λογιστικά, που θα διευκολύνει το έργο των μικρών και μεσών επιχειρήσεων. Η ίδια η Κομισιόν καταθέτει έγγραφο για τις εξαιρέσεις μικροεπιχειρήσεων από διοικητικά βάρη και έχουν και νέους τρόπους για να ελέγχουν την επάρκεια της νομοθεσίας σε όλη την δέσμη των ευρωπαϊκών νομοθετημάτων και για να εντοπίσουν για το μέλλον 10 τομείς όπου μπορούν να μειώσουν τις γραφειοκρατικές ρυθμίσεις. Ε, ανοίγονται λοιπόν εκεί κάποιες ευκαιρίες. Η κυρία Τόγια είπε ότι πρέπει να έχουμε υπόψη το γεγονός ότι οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις έχουν μικρή γραφειοκρατική ικανότητα και εκεί μπορεί να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα κολλήματα. Αυτό είναι θέμα εθνικού επίπεδου. Με τις ανεπίσημες επαφές μας θα εξετάσουμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές για να δοθεί καλύτερη πρόσβαση στις μικρές και μεσές επιχειρήσεις σε προγράμματα που είναι ειδικά για αυτές. Για μικρές και μεσές επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν το managing time που έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή την ε, διοικητική ικανότητα. Έτσι λοιπόν πρέπει ε, να τονιστεί και ο θεσμός των first, shop, των first stop shop και άλλων πρωτοβουλειών, μικροπιστώσεις και ούτω καθεξής. Διαφορετική είναι η έμφαση που δίνει στην προστασία δεδομένων ο Σον Κέλλη και η κυρία Άντερς Ντότερ. Εδώ βέβαια πρέπει να επιτευχθεί μια ευαίσθητη ισορροπία όσον αφορά την προστασία της προσωπικής σφαίρας, των χρηστών, τα διάφορα θέματα copyright των ατόμων και ούτω καθεξής Χρειάζεται ωστόσο μια δόμηση μιας στέρεας ψηφιακής οικονομίας. Όμως, αν πετύχουμε σωστή ισορροπία, ανοίγονται πάρα πολλέ ευκαιρίες. Γνωρίζω ότι γίνεται πολλή δουλειά και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εξασφαλιστεί ακριβώς αυτή η ορθή ισορροπία. Για την κυρία Άντερς Μπαρέα, που μίλησε για την δημιουργία απασχόλησης και ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα. Βέβαια, χρειάζεται να συνεξετάσουμε όλα τα δεδομένα. Υπάρχουν ενθαρρυντικά προγράμματα στις μικροπιστώσεις αλλά και σε άλλες μορφές χρηματοδότησης. Επίσης το εμπόριο, η εκμετάλλευση των ευκαιριών της ενιαίας αγοράς, αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της εκπαίδευσης, η λεγόμενη Youth Guarantee. Όλα αυτά είναι προγράμματα που ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προωθήσουμε σημαντικά, ανοίγοντας έτσι ευκαιρίες για περισσότερη απασχόληση, για εξασφάλιση πρόσβασης. Η κυρία Χίπνερ μίλησε εν παρόδο για ταχύτερες οδούς προς την εξασφάλιση ευρεσιτεχνιών. Αυτά έχουμε να τα συζητήσουμε στο Συμβούλιο του Φεβρουαρίου για να μειωθεί το κόστος των ευρεσιτεχνιών για μικρές και μεσές επιχειρήσεις με την έννοια ότι δεν θα χρειάζεται να υποβάλουν αιτήσει για διπλώματα ευρεσιτεχνιών σε όλες τις χώρες με ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να επιφέρουμε κάποιες βελτιώσεις. Αυτά ήταν τα θέματα που έχουν άμεση σχέση με το δικό μου χαρτοφυλάκιο και βέβαια περισσότερα έχει να πει ο Σον, μιας και τα θέματα του είναι για τον ορίζοντα 2020. Ευχαριστώ, Ρίτσαρντ. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω γενικά ότι καλύφθηκαν πάρα πολλά θέματα εδώ, τις ερωτήσεις και οποιαδήποτε εταιρεία οποιαδήποτε χώρα πρέπει να βασιστεί στην ε, δική της εμπειρία, βλέποντας τη δική της ιστορική και πολιτική προοπτική. Και στα πλαίσια του ορίζοντος 2020 πρέπει να προδεύσουν διάφοροι φάκελοι στους οποίους έχουμε μεγάλη εμπειρία εμείς στην Ιρλανδία. Δηλαδή, να δημιουργήσουμε σιγά σιγά τις συνθήκες για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Και ξέρουμε εδώ ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη-μέλη. Έχουμε προβλέψει να οργανώσουμε διασκέψεις, έχουμε κοινέ συνεδριάσεις τις συμπεράσματα των οποίων θα παρουσιάσουμε το Μάιο στο Συμβούλιο και μας απασχολεί πάρα πολύ το θέμα της προόδου όλου του φακέλου της έρευνας στην Ευρώπη, διότι πιστεύουμε ότι είναι πρωταρχικής σημασίας για να μπορέσει παγκοσμίως να είναι η Ευρώπη ανταγωνιστική. Και πιστεύουμε ότι η πρόοδο σε όλους αυτούς τους σχετικούς ε, φακέλου. Δεν ξέρουμε πόσο μακριά θα πάμε, αλλά ε, φιλοδοξούμε να προχωρήσουμε πολύ ώστε να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί διεθνώς. Τώρα, είπα ότι προσπαθούμε να προχωρήσουμε στα πλαίσια της ε, νομοθεσίας και των ε, κανονισμών και στα πλαίσια των μικρομε... το τι μπορούμε να κάνουμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα πλαίσια του προγράμματος ε, που αφορά τους κανονισμούς που θα παρουσιαστούν, κυρίως στα πλαίσια του ε, πολιετούς χρημα... Ε, δημοσιονομικού πλαισίου. Τα θέματα των κονδυλίων είναι σημαντικά, έχουν σχέση με το πολιετές αυτό πλαίσιο. Για όλους τους φακέλους όπως και για το πρόγραμμα Horizon 2020. Είναι σημαντικό σε θέματα απλοποίησης όπως αναφέρθηκε και δεσμεύσεις υπέρ των ΜΜΕ να ενεργήσουμε από κοινού. Ξέρουμε ότι είναι συμπληρωματικές οι θέσεις μας, διότι προτείνουμε να αυξηθεί κατά 20% η χρηματοδότηση που προβλέπεται. Και βεβαίως και οι δύο χαιρετίζουμε στα πλαίσια του ορίζοντος 2020 την απλοποίηση. και να μπορέσουν να συμμετέχουν πιο εύκολα οι μιμιέ. Αυτό είναι θέμα το οποίο θέλουμε να συζητήσουμε μέσω της διαδικασίας του διαλόγου των τριών θεσμικών οργάνων ώστε όλοι να έχουν ίσους όρους πρόσβασης. Επειδή οι θέσεις μας λοιπόν είναι παρεμφερείς πιστεύουμε ότι θα υπάρξει πρόοδος. Τώρα, για ειδικά θέματα τα οποία αναφέρθηκαν για την πολιτική βιομηχανίας και πόσο σημαντική είναι η βιομηχανία διαστήματος στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό πρότυπο της, του οργανισμού του Ευρωπαϊκού είναι πολύ καλό και θα πρέπει εδώ να δημιουργηθούν νέες ε, δυνατότητες της ε, βιομηχανίας μέσα της Ευρώπης για την αγορά. Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την πολιτική που θα ακολουθηθεί αναμένεται με ενδιαφέρον, διότι όπως είπε ο κύριος Κέλλη, ότι κάνουμε είναι κάτι το οποίο αφορά όλη την Ευρώπη. Και θα πρέπει εμείς ε, να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και να διευκολύνουμε και τη συμμετοχή των ΜΜΕ σε θέματα βιομηχανίας του διαστήματος στην Ευρώπη. Γενικά λοιπόν προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα διευκολύνουμε την συμμετοχή, ότι θα προοδεύσουμε στην υλοποίηση των στόχων, τα 20 τουλάχιστον 100%, προσπαθούμε να επιτύχουμε την ε, διευ... απλοποίηση των διαδικασιών και οι διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του ορίζοντος 2020 του προγράμματος αυτού ελπίζω να μπορέσουν να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της δικής, του δικού μας εξαμήνου. Και αναμένονται οι διαπραγματεύσεις και η ολοκλήρωση του στα πλαίσια του πλαισίου, του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και το πρόγραμμα Horizon 2020 θα αποτελέσει τελικά, ελπίζουμε, ένα μέσο δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης για όλη την Ευρώπη. Ο στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να ολοκληρώσουμε τις σχετικές διαπραγματεύσεις. So that's, broadly it. Uh, Αυτά ήθελα να πω κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι κάλυψα τα ερωτήσεις που αφορούσαν τον τριμερή διάλογο, του στόχους των ΜΜΕ και το πρόγραμμα Horizon 2020 καθώς και το πλαίσιο δημοσιονομικού πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους Υπουργούς ε, για την παρουσία τους, ε, για την προθυμία τους. Ε, αλλά και για τις που ανέλαβαν ενώπιόν μας. Ε, τους ευχαριστούμε για τις προσκλήσει ε, που μας ε, έκαναν και ελπίζω και νομίζω πως αυτό είναι επιθυμία όλων μας ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία πλήρω των τριμερών διαλόγων διότι έχουμε πολλούς μπροστά μας. Σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά έξω ονόματος των συναδέλφων και σας υπενθυμίζω ότι αύριο το πρωί σε 9 θα τα ξαναπούμε εδώ. <laughs> Merci beaucoup.